Άρχεται η συνεδρίαση. Καλημέρα προς όλους. Λοιπόν, ξεκινούμε με μία ανακοίνωση. Η κυρία Collins εγκαταλείπει την ομάδα ENF και προσχωρεί στην ομάδα EFTD από τις 17 Απριλίου 2019. Επίσης, η κυρία η Ελίζαμπέτα Γκαντίνη εγκαταλείπει το, την ομάδα του ΕΛΚΑ και προσχωρεί στους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές από τις 17 Απριλίου 2019. Ξεκινούμε με την ημερήσια διάταξη. Έκθεση μπάλας για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Το λόγο έχει ο εισηγητής κ. Μπάλας για 4 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Δεκέμβριο του 2016 η αναθεώρηση του κανονισμού 883 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας υποβλήθηκε ως πρόταση από την Επιτροπή. Υπάρχει σήμερα μια ανάγκη όντως να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον υπάρχει το εξής παράδοξο. Έχουμε μια αγορά η οποία επιτρέπει την ελευθερία κυκλοφορίας, αλλά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης εξαιρετικά διαφορετικά, άρα καταστάσεις τροτότητας των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την προστασία και την μεταφορά των δικαιωμάτων αυτών. Αυτό είναι το στόχος του, της πρότασης Επιτροπής. Συνεργαστήκαμε για πάνω από ένα έτος στο Κοινοβούλιο και καταλήξαμε νομίζω σε τρεις μεγάλες ε, και σημαντικές πρόοδους. Πρώτον, ουσιαστικό. Ενίσχυση της εφαρμοστέας ε, νομοθεσίας, δηλαδή ε, επίγνωση της νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε ένα εργαζόμενο, ένα αποσπασμένο για παράδειγμα. Για ένα ουσιαστικό στοιχείο στο σημείο αυτό είναι να εξασφαλίσουμε ότι ένας εργαζόμενος είναι πραγματικά συνδεδεμένος με ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, άρα απολάβει όλων των δικαιωμάτων. Γι' αυτό προτείναμε να υπάρξει μία περίοδος τριών μηνών προγενέστερης εργασίας πριν ένας εργαζόμενος αποστελεί σε άλλη χώρα για να εξασφαλίσουμε την σύνδεση μεταξύ του εργαζόμενου και του συστήματος ε, και της ένταξη ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό για να αποφύγουμε τη... τις περιπτώσεις απάτης που γνωρίζουμε. Ομοίως, μια άλλη πρόταση που υιοθετήσαμε είναι η αλλαγή, η προγενέστερη αλλαγή από μια επιχείρηση της αποστολή ενό εργαζομένου σε άλλη χώρα. Είναι ουσιαστικό αυτό σήμερα, διότι όπως γνωρίζουμε, ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων που αποστέλλονται σε τρίτε χώρες δεν είναι καν γνωστοί στις χώρε αυτέ, γιατί ορισμένε εθνικέ νομοθεσίε ιδίω δέχονται ότι ε, εντεύθεν ε, για, για μια περίοδο μικρότερη από ένα χι διάστημα δεν χρειάζεται κανένα έγγραφο, άρα δεν μπορεί να γίνει κανένα έλεγχο για το συγκεκριμένο εργαζόμενο. Εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσβολή τη αξιοπρέπεια του εργαζομένου, τη ασφάλειά του και των δικαιωμάτων του εργαζομένου να εντάσσεται σε ένα σύστημα κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πρόταση κοινοποίησης. Επίσης, βελτιώνουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, κάτι που ζήτησε το Κοινοβούλιο, ιδίω με ένα ε, πρωτότυπο σύστημα που συνδέει που επιβάλλει δέσμευση στα κράτη-μέλη με κατάθεση εγγύσεων και την ελευθερία κυκλοφορίας, διότι παρέχει μια μεγάλη ευελιξία στον εργαζόμενο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να περάσει από το ένα σύνορο στο άλλο μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, ε, έξι μήνες εξαγωγής. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποιος που είναι δύο χρόνια σε μια χώρα φεύγει από μια χώρα και έχει μόνο τρία, τρεις μήνες δικαιώματος επιδόματος σε επίδομα ενεργείας. Έξι μήνες είναι σαφώς καλύτερο. Κάτι που μπορεί να φανταστείτε ότι είναι σημαντικό ιδίω για τους διασυνοριακούς, για τους μεθοριακούς εργαζομένους. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόοδο. Να πω τα εξής προς την δεξιά, τις δεξιές, αλλά όχι μόνο. Μην πιστεύετε ότι μιμούμενοι τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό θα απαντήσετε στους εθνικισμούς και τους λαϊκισμούς. Μερικές φορές το, είναι τέτοιο παραδοξό που ορισμένοι εθνικοί τεστές έγιναν πιο φρόνιμη από ότι σε εσά τα συστήματα συντονισμού των, κοινωνικών, ε, των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης. Μην εμποδίζετε λοιπόν μόνιμα τι συζητήσει. Αφήστε του βουλευτέ σα να ψηφίσουν ελεύθερα, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή θέση ενώπιον εν ώψη τη επόμενη θητεία. Α ψηφίσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ανάγνωση και ω προ το μέλλον να πω προ την Επίτροπο, την ευχαριστώ για το έργο που κατέβαλε, με πλήρη συμφωνία, ούτω ώστε ο συντονιστικό κανονισμό να αναθεωρείται με απλή πλειοψηφία στο Συμβούλιο για να μην υπάρχει παρεμπόδιση που διαπιστώνουμε πολύ πρόσφατα, δύο εβδομάδες πριν, αποτελεί μια μεγάλη πρόοδο για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους που επιτέλους θα μπορέσουν να προστατευθούν εις βάρος των εθνικών ευρωριζών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή. Το λόγο έχει τώρα η Επίτροπος κυρία Τέισεν, την οποία ευχαριστώ για την παρουσία της εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Συγητά, αξιότιμα μέλη, είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για να συζητήσουμε το θέμα του συντονισμού των ε, κοινωνικών συστημάτων, συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Ε, προτείνουμε μια, ένα καινούριο εξυγχρονισμό 15 χρόνια μετά τον προηγούμενο κανονισμό 883, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις ε, σε ό,τι αφορά τις παροχές ανεργίας, τις παραοικογενειακές ε, παροχές, τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζόμενων κλπ. Υιοθετήσαμε την πρότασή μας πριν από δύο χρόνια για να εξασφαλίσουμε την δικαιοσύνη στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην εσωτερική αγορά και των εργαζομένων. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλα, στον εισηγητή, καθώ επίση και τα πολλά μέλη του Κοινοβουλίου που πραγματικά επένδυσαν χρόνο και ενέργεια σε αυτό το θέμα για να βελτιωθούν οι προτάσει μα προ όφελο των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των πολιτών μα. Η διευκόλυνση ε, των ε, οικογενειακών ε, παροχών και αδειών, η διευκόλυνση, η, η αποσαφήνιση του καθεστώτος της ε, μακροχρόνιας περίθαλψης κλπ. είναι παραδείγματα του πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των πολιτών. Για μένα, πάντοτε ήταν απαραίτητος ο συντονισμός των συστημάτων ε, ε, κοινωνικής ασφάλισης με κανόνες που να είναι σαφείς, ε, δίκαιοι και να και εφαρμόσιμοι. Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την συνεχή στήριξη της εσωτερικής μας αγοράς. Δικαιοσύνη σημαίνει ότι οι κανόνες θα είναι ισο, ίσοι ίδιοι για όλους και δεν θα έχουν σχεδιαστεί για να ωφελούν ε, μία ομάδα εις βάρος κάποιας άλλης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα και του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους ε, μέλους προορισμού. Επίσης, η δικαιοσύνη σημαίνει ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα μετακινούνται σε άλλη χώρα υπό Σωστέ συνθήκε, λαμβάνοντα υπόψη τα ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα των φορολογουμένων, αλλά και τι ανάγκε, τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης να είναι ε, βιώσιμα. Επίσης, δικαιοσύνη σημαίνει καινούριε ευκαιρίε για όλες τις ε, επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους ε, που θα πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες όλης της Ευρώπης. Επίσης δικαιοσύνη σημαίνει το να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των καταχρήσεων και τη απάτη. Αυτέ είναι οι αρχέ πάνω στι οποίε έχουμε βασίσει τι προτάσει μα. Είναι και στόχοι, άλλωστε, που, μας, ε, ε, που ήταν ο γνώμονάς μας ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η προσωρινή συμφωνία στην οποία φτάσαμε κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου δεν επιβεβαιώθηκε, διότι δεν εξασφαλίστηκε επαρκής πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών. Όμω πιστεύω ότι ο συμβασμός τον οποίο πετύχαμε θα πρέπει να μας εμπνεύσει για το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγητά, κύριε Σιγητές, αγαπητοί ευρωβουλευτές, αυτό το Κοινοβούλιο έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να ε, συμφωνήσει ε, να βρει μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και να ανοίξει ένα ορίζοντα για πρόοδο σε αυτό το θέμα στο μέλλον. Ε, βασίζομαι στην επικοδομητική σας προσέγγιση και στο ότι ε, μοιραζόμαστε την επιθυμία να επωφεληθούμε τη ευκαιρία προ όφελο των επιχειρήσεων, των πολιτών μα ε, και γενικά τη Ευρω... Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Α ακούσουμε τι απόψει των πολιτικών ομάδων τώρα. Στην πρώτη αυτή φάση δεν γίνονται δεκτέ οι μπλε Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σούλτσε, 1,5 λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επιτροπέ. Κυρίε και κύριοι, από πλευρά μου, ο συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς νόμους ε, και πραγματικά προώθησε την Ευρώπη και ουσιαστικά ρυθμίζουμε την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, μία από τις βασικές ιδέες της ΕΕ. Αγαπητοί συνάδελφοι, για τη σημαντική αυτή νομοθεσία θεωρώ ότι δεν δαπανίσαμε επαρκή χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επέβαλε καθυστερημένα ουσιαστικά την πρόταση της και σε όλη την Ευρώπη είναι ουσιαστικά δύσκολο να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μεγάλη χρονική πίεση για την ε, ψηφοφορία στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή μα και για του τρομερεί διαλόγου. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Άρα δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να, αποτελε... για να βρούμε ένα καλό ε, αποτέλεσμα στο οποίο θα συμφωνήσει και το Συμβούλιο. Έχουμε και ανάγκη για συντονισμό σε άλλα θέματα, σε ό,τι αφορά την απόσπαση, τα ταξίδια, τα επαγγελματικά για να υπάρχουν βράχοι πρόθεσμες ε, αποσπάσεις. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μας απασχολούν. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την απόσπαση και σε ό,τι αφορά την διακοπή της απόσπασης. Μια καλή ιδέα η οποία όμως δύσκολα εφαρμόζεται ψηφιακά. Για παράδειγμα, όταν είναι κάποιος δάσκαλος και πηγαίνει σε ένα άλλο σχολείο, είναι απόσπαση ή όχι. Αναφέραμε το θέμα των εξαγωγών, το θέμα της επιλογής συστημάτων, το οποίο ενδεχομένως θα πλήξει τις διασυνοριακές ε, περιοχές. Στον τριμερή διάλογο το πετύχαμε, αλλά δεν ψηφίζουμε το αποτέλεσμα του τρομερού διάλογου. Χρειαζόμαστε πιο πάρα πολύ χρόνο, θεωρώ, για να το κοιτάξουμε αυτό στο νέο κοινοβούλιο και το η ομάδα του ΕΛΚ θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα μετά τις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ κυρία Ιονγκέριους για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε μπροστά μας ε, ένα μεγάλο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά ε, θετικά στοιχεία αλλά και αρνητικά στοιχεία και τελικά θα αναγκαστούμε να ψηφίσουμε κατά της ε, πρόταση αυτή, όχι κατά τη ιδέα, αλλά κατά τη υλοποίηση. Στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο μεγάλε υποθέσει οργανωμένη απάτη σε ό,τι αφορά τα επιδόματα ανεργία. Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι όλοι συνεισφέρουν και κανεί δεν λαμβάνει ε, επιδόματα χωρί να έχει δικαίωμα. Γιατί ουσιαστικά με τι συνεισφορέ του το πληρώνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Και στην πρόταση ουσιαστικά. Ε, με την πρόταση αυτή σταματάει να υπάρχει υποχρέωση αναζήτηση εργασία στην αγορά εργασία. Και σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές επιδομάτων έχουμε πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την ε, παράταση ε, συμβάσεων κλπ. Κάτι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους από την ανεργία, γιατί για μας η αλληλεγγύη του συστήματος είναι η πρώτη φροντίδα. Και δεν θεωρώ ότι εγγυαόμαστε αυτό με την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το ECR τώρα έχουμε την κυρία Στίβενς για μισή λεπτό. Και για σας. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Όλοι μας συμφωνούμε ότι η κοινωνική απάτη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στεναρά. Οι κοινωνικές επιθεωρήσεις όλων των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται, για παράδειγμα, πολύ πιο ε, επαρκώς. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη προθεσμία εργασίας πριν οι εργαζόμενοι από άλλες χώρες μπορούν να ζητήσουν επιτόμητα ανεργία. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ε, οι εργαζόμενοι που δεν είναι από το Βέλγιο θα πρέπει πρώτα να συνεισφέρουν στην ε, κοινωνική ασφάλεια του Βελγίου προτού έχουν δικαίωμα ε, επιδομάτων ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον τρει μήνε να ζητούνται ω περίοδο ε, συνεισφορά προτού ζητάει ο εργαζόμενο επιδόματα. Έξι μήνε θα ήταν ακόμα καλύτερο. Κάποιοι θα θέλαν ο εργαζόμενο να έχει δικαίωμα σε επίδομα ανεργία από την πρώτη ημέρα. Αυτό πραγματικά είναι καθαρή ανοησία, γιατί υπονομεύει τη βάση τη κοινωνική μα ασφάλιση. Επίση, η αριστερά θέλει οι άνθρωποι που ψάχνουν δουλειά να έχουν δικαίωμα να πάρουν μαζί του ε, το επίδομα ανεργία αν μετακομίσουν στη χώρα προέλευσή του. Αλλά ουσιαστικά αυτό ακυρώνει οποιοδήποτε έλεγχο. Και αυτό ουσιαστικά προωθεί την απάτη. Γιατί οι στατιστικέ καταδεικνύουν ότι μεγάλο αριθμό ε, ατόμων που επιστρέφει στην χώρα του, στην πατρίδα του, δεν βρίσκει δουλειά του τρει πρώτου μήνε. Και γιατί να βρουν δουλειά άλλωστε, αφού με το βελγικό επίδομα ανεργία μπορεί κανεί να ζήσει πολύ, πολύ άνετα σε μια χώρα τη Ανατολική Ευρώπη. Η Φλάνδρα είναι μια οικονομία η οποία προσανατολίζεται στι εξαγωγέ, αλλά η κοινωνική μα πρόνοια δεν είναι προϊόν εξαγωγή. Με άλλα λόγια, χωρί συνεισφορέ δεν έχει και παροχέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για τους ελεύθερου. η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Είμαστε νομοθέτες και άρα έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίζουμε ότι οποιοδήποτε νομοθετικό κείμενο υποστηρίζουμε θα βελτιώσει την φυστάμενη κατάσταση, θα εντοπίσει και θα λύσει προβλήματα. Θα συμβάλλει στην ελεύθερη και δίκαιη μετακίνηση των εργαζομένων και θα εξασφαλίσει εμπιστοσύνη, ασφάλεια δικαίου και κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και ισότιμη αντιμετώπιση όλων. Αυτά είναι τα ορόσημα μας στους φιλελεύθερους. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής είναι μια αξιοπρεπής προσπάθεια να πετύχει ένα βελτιωμένο καθεστώς. Το σχέδιο συμφωνίας στον Τρίλογο έχει μια σειρά θετικών στοιχείων που, δεν, που υπερστήριξε το Συμβούλιο. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία στη σημερινή έκθεση για τα οικογενειακά επιδόματα, τη μακροχρόνια ε, παροχή ε, επιδομάτων υγείας. Ωστόσο, οι τροπολογίες στο άρθρο 13 που θα μπορούσαν να ε, βελτιώσουν θεωρητικά την κατάσταση των οδηγών θα οδηγήσει σε πολύ κακές συνέπειες υπάγοντας τους οδηγούς σε διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υποβάλλουμε μια σχετική τροπολογία. Δεν συμφωνούμε ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι μπορεί να επιλέξουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα χρησιμοποιήσουν, διότι αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια στα κράτη-μέλη και θα υπονομεύσει το κοινωνικό συμβόλο μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών εργαζομένων. Δεν υποστηρίζουμε την ανομαλία που θα δημιουργήσει μεταξύ ε, μεταξύ διασωνεριακών και εθνικών εργαζομένων. Μπορούμε να δεχθούμε κάποιες τροπολογίες και να υποστηρίξουμε το νομοθετικό κείμενο συνολικά. Αν γίνουν δεκτές οι τροπολογίες μας, αν όχι, δεν θεωρούμε ότι θα δώσει ισορροπημένη ισορροπημένο αποτέλεσμα. Θέλω να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους όδης εισηγητής γιατί δούλεψαν για το φάκελο αυτό με, με, με προσπάθεια. Μπορεί να μην συμφωνήσαμε παντού αλλά δουλέψαμε όλοι μαζί. Η κυρία Τζίμερ για την ομάδα της Γκούες για δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, μου φαίνεται μετά από αυτά που άκουσα ότι ένα τμήμα των συναδέλφων εδώ στο Κοινοβούλιο δεν κατανοούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν τη βασική αρχή της συντονισμού των κοινωνικών ασφαλίσεων. Μιλάμε για δικαιώματα τα οποία έχουν αποκτηθεί σε ένα κράτο μέλο να αναγνωριστούν σε ένα άλλο κράτο μέλο. Τίποτα παραπάνω. Όποιο λέει ότι μπορεί κανεί να έχει δικαίωμα και να αποκτήσει δικαίωμα εφόσον έχει συνεισφέρει στο άλλο σύστημα, ουσιαστικά αγνοεί και υπονομεύει αυτή την αρχή. Να σταματήσουμε να μιλάμε για μια ένωση γεωνική πρόνοια, λοιπόν. Σα παρακαλώ, επιτέλου, ε, ομολογήστε. Θέλετε να κάνετε με να αποτρέψετε αυτή τη συζήτηση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Είναι μη δημοκρατικό αυτό, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, αλλά να μην κάνουμε τη συζήτηση καν και να μην γίνει ψηφοφορία. Στην τρέχουσα θετία αυτό δεν έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτή η επιλεκτική εμ, επιλογή εμ, κοινωνικών συστημάτων καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όλοι να έχουν κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και η πλειοψηφία της Επιτροπής Απασχόλησης υπερψήφισε μια προοδευτική πρόταση, την οποία και συζητούμε. Θα ψηφιστεί λοιπόν αυτή η πρόταση. Εμείς ως αριστερά, ως Λίνκε, ξέρουμε ποια είναι η τοποθέτησή μας σε ό,τι αφορά και τους έξι μήνες υπερψηφίζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κλείσουν τα κενά που δημιουργούνται στην ε, οδηγία για την απόσπαση. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός, αλλά Είμαστε κατά της απόπειρας κάποιων συντηρητικών και ακροδεξιών να προσπαθήσουν να περάσουν προσαρμογή και διόρθωση του επιδομάτως τέκνων. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος ο οποίος εργάζεται στη Γερμανία από την Ανατολική Ευρώπη να έχει λιγότερα επιδόματα τέκνου, γιατί τα παιδιά του είναι στην Πολωνία, για παράδειγμα. Αυτό είναι κοινωνική αδικία για άτομα τα οποία έχουν πληρώσει τι συνεισφορέ του και θέλουν να φροντίσουν τα παιδιά του που είναι στην πατρίδα του. Θέλουμε λοιπόν να σταματήσουμε να το συζητάμε το θέμα αυτό. Το θέμα επίση τη κοινωνική ισότητα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Όλου του Ευρωπαίου πολίτε θα πρέπει να προσπιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανεί δεν μπορεί να είναι δεύτερη κατηγορία πολίτη. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για τα επιδόματα ανεργία όταν έχει πληρώσει κανεί ε, τι συνεισφορέ του σε ένα κράτο, θα πρέπει να γνωρίζεται αυτό σε άλλο κράτο. Και υπάρχει ένα βασικό κανόνα ε, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Θα πρέπει ω Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσουμε, τελευταία πρόταση, σε όλε τι χώρε οι πολίτε να έχουν δικαίωμα στα συστήματα κοινωνική ασφάλιση. Ευχαριστώ. Για η Λάμπερτ, δυόμιση λεπτά να σεβόμαστε το χρόνο γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίες σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ε, έφτασα πριν από 20 χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο, ο πρώτος φάκελος στον οποίο εργάστηκα ήταν η συνολική αναθεώρηση της συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Και ψηφίσαμε εκείνη την συμφωνία που έγινε κανονισμός με τον αριθμό 883 ε, στην τελευταία ολομέλεια εκείνη τη θητεία μα. Ελπίζα ε, ότι θα είχαμε καταλήξει μια παρόμοια συμφωνία με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση αυτού του κανονισμού. Δυστυχώς όμως εξαιτία του, του διχασμού στο Συμβούλιο δεν τα καταφέραμε. Αυτό το θέμα ε, έγινε ένα μείγμα μικροσυμφερόντων, εθνικών μικροσυμφερόντων, ε, ανθρώπων ε, που προσπαθούν να λύσουν μέσω αυτού του κανονισμού πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την ουσία του. Κατά την άποψη της ομάδας μας, το, αυτό που πρέπει να έχουμε στο κέντρο της σκέψης μας θα πρέπει να είναι οι πολίτες, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, τα μέλη των οικογενειών τους κλπ ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται. Χαιρόμαστε που έχει συμπεριληφθεί η μακροχρόνια περίθαλψη. Όμως, ε, σημείο φετηρία μας είναι ότι η πλειοψηφία των, των πολιτών και η επιχειρηματίες είναι, ε, επιθυμούν να είναι νόμιμοι, να μην κάνουν απάτες και παρανομίες. Οπότε είναι χρήσιμο οι να είναι απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους, ευέλικτοι έτσι ώστε να τους βοηθάνε στην καθημερινότητά τους. Επίσης θα χρησιμεύε οι διοικητικέ δομές να είναι αποτελεσματικές και να μπορούν να, απαντήσουν, να απαντούν γρήγορα και να μην δρούν ως γραφειοκρατικό εμπόδιο. Εν γέννη, συμφωνούμε με την έκθεση της Επιτροπής. Η μόνη τροπολογία, η 197 την οποία ε, προβάλαμε, ε, ε, έχει σχέση με, την, με τους ανθρώπους που ε, εργάζονται, που κάνουν πολλά επαγγελματικά ταξίδια, να μην χρειάζονται να ε, ζητούν συνεχώς ε, βεβαίωση κάθε τόσο για κάθε τους ταξίδι. Οι βεβαίωση να διαρκούν τρει μήνες. Επίσης δεν στηρίζουμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών επιδομάτων. Αυτό το μέτρο δεν θα, ήταν, δεν θα είχε επαρκές όφελο σε σχέση με το κόστος του. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση ε, ενισχύει τις δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου των κρατών μελών. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσαν ε, να υιοθετήσουν έκτακτα διμερή μέτρα αν χρειαζόταν, αν υπάρχει ένα διμερές πρόβλημα. Οπότε η πρόταση αυτή βρίσκεται σε μια σταθερή βάση και αποτελεί πολύ καλή βάση για διαπραγμάτευση στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ ο κύριος Σούλτσε ε, θέλει κάτι, αλλά δεν είναι εδώ. Πούντος. Ζητήσατε το λόγο για, για ποιο λόγο όμως, παρακαλώ. Πρόεδρε, για ένα δεδικαστικό θέμα θα ήθελα να μιλήσω. Αυτά τα 10 λεπτά που καθυστέρησαν, ξεκίνησαν τη συζήτηση 10 λεπτά αργότερα. Δεν ε, έχω δικαίωμα για μπλε κάρτα και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τσίμερα αν είχα μπλε κάρτα. Τι είδου κόλπα θεωρεί ότι ε, ε, κάνουμε εμείς ως δεξιά για να υποβάλουμε τροπολογίες. Δεν είναι κόλπο αυτό και αν είχατε έρθει στην ώρα σας θα μπορούσα να κάνω την ερώτησή μου στα πλαίσια της μπλε κάρτας. Μα δεν κατάλαβα. Τι θέλετε. Μισό λεπτό. Για την ομάδα EFDD. ο κύριος Κόμπουρν έχει το λόγο για 3,5 λεπτά. Λείπει. Επόμενος, για την ε, ομάδα ENF, η κυρία Μελέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το κείμενο αυτό, η ομάδα μας έχει μία στάση αναμονής και περισυλλογής. Διότι αν το κείμενο αυτό που είναι πολύ παλιό και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια της συνεργασίας όπως την εμείς αντιλαμβαζόμαστε στα πλαίσια μιας συμμαχίας ευρωπαϊκών εθνών. Το κείμενο το τωρινό βελτιώνει κάποια πράγματα την ακόψή μας ιδίως ότι αφορά την ασφάλεια που παρέχεται στους μεθοδιακούς εργαζομένους οι και στα παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται σε άλλη χώρα. Γιατί και εμείς θέλουμε το απόλυτο δόγμα της χώρας που εισπράττει τις εισφορές να είναι η χώρα που καταβάλει παροχές. Αντίθετα, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις προς το κείμενο. Ένα τεράστιο πρόβλημα που διαπιστώνουμε αφορά τον καθορισμό της περιμέτρου της ε, μακροχρόνιας ασθένειας. Στην ε, Γαλλία καλύπτει το 70% του προϋπολογισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές χώρες. Επίσης, δεν ε, συμφωνούμε με το γεγονός ότι το κείμενο του εισηγητή επιβάλλει σβήνει την νόμιμη υποχρέωση παραμονής του δικαιούχου και στηριζόμαστε πλέον μόνο σε νομολογία που μπορεί και αυτή να ερμηνευθεί. Επίσης μας ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Α, υπάρχει αντιπολίτευση και άρνη σε κάποια σημεία, ιδίω η δεξιά και δεν επιτρέπει και γι' αυτό δεν οδήγησε σε αποτέλεσμα ο τρίλογος, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε βεβαιότητα για την πρώτερη ε, αδειοδότηση. Για να μπορέσει το κείμενο αυτό να περάσει πρέπει να περιλάβει οπωσδήποτε την ε, μια απαγόρευση πιθανών απατών ιδίως μέσω της πρώτερης ε, αδειοδότησης. Ευχαριστώ. Σόσνιατς από τους μη για ένα λεπτό. Κυρίε και κάθε φορά που παίρνουμε κάτι από κάποιον ή να το δώσουμε σε κάποιον άλλον, ε, συνήθω μα οδηγεί στο να παίρνουμε από αυτού που δουλεύουν για να δίνουμε σε αυτού που δεν δουλεύουν. Αυτό είναι ανήθικο. Ε, μα ζητούν αλληλεγγύη μεταξύ αυτών που δουλεύουν και αυτών που δεν δουλεύουν. Αυτό οδηγεί σε απίστευτη γραφειοκρατία και άχθος. Μη λέτε ότι θέλετε να εξασφαλίσετε την ελευθερία κυκλοφορίας ενώ ταυτόχρονα επιτρέπετε ε, αδειοδοτήσεις, έρευνες, ε, επιθεωρήσεις κλπ. Ε, αν τα ε, οι παροχές είναι πρόβλημα, ας καταργήσουμε τις παροχές. Αν η απάτη είναι πρόβλημα, ας καταργήσουμε τις παροχές. Ε, η αριστερά θέλει να προωθήσει ένα πολύ επίμαχο θέμα, γνωρίζοντας ότι ο λαός έχει βαρεθεί πια. Δεν θέλουμε πια σοσιαλιστικά πειράματα. Ευχαριστώ. Ωραία, ακούσαμε τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους. Ξεκινάει γενικότερη συζήτηση. Κάζα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθεσία που θα επηρεάσει όλα τα κράτη-μέλη και την ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ένωση. Οι προτάσεις αλλαγών είναι πολλές και καλύπτουν μέτρα για άνεργους, πρόσβαση σε μη ενεργούς ε, οικονομικά εργαζόμενους, ε, αποσπασμένους εργαζόμενους κλπ. Η διαφοροποίηση των εθνικών νομοθεσιών έχει δημιουργήσει μια σειρά ερωτημάτων, αλλά χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μια σειρά προσωρινών ε, συμφωνιών θέτουν σε κίνδυνο την σαφήνεια του κειμένου, ιδίω και λόγω της έλλειψης πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Δεν πρέπει να κάνουμε λοιπόν οποιαδήποτε ε, λάθη. Κάθε αλλαγή πρέπει να βελτιώνει την κατάσταση και να μην δημιουργεί εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και στους εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους. Ξέρω ότι υπάρχουν μια σειρά τροπολογιών επιτάπητος. Στις ψηφοφορίες αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τροπολογίες βελτιώνουν την νομοθεσία και είναι θετικές για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους κοιόδης εισηγητέ. Δεν, συμφωνήσαμε, δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά δουλέψαμε καλά γιατί προσπαθώντας να βρούμε κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να μας βρει σύμφωνο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέσο. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, είναι σίγουρο ότι η επικαιροποίηση των κανόνων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και την πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους κοινού, μετακινούμενους εργαζομένους που αυξάνονται στην Ευρώπη είναι βασική προϋπόθεση για να έχουμε μια πιο κοινωνική και συμπεριλαμβάνουσα Ευρώπη ο κατακαιρματισμός των εθνικών συστημάτων, συστημάτων ασφάλισης έχετε, πάει εις βάρος των στόχων αυτών. Ε, ο συντονισμός, ακόμα και ο συντονισμός θα μπορούσε να αποτελέσει μια, ένα μεγάλο βήμα μπρος για την νομοθετική σαφήνεια. Ωστόσο, για κάποια ζητήματα που θεωρούμε σημαντικά, όπως ε, αυτά που αφορούν τους μεθοδιακούς εργαζομένους, τους διεθνικούς εργαζομένους που μπορούν να αποφασίσουν πού θα λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας και που είναι ευάλωτοι εργαζόμενοι που πρέπει να, να προστατευτούν ενώ ένα άλλο σημείο σύνθετο έχει να κάνει με τον τρόπο και τον τόπο όπου θα λαμβάνονται τα επιδόματα ανεργίας για όποιον αναζητά εργασία σε μια άλλη χώρα. Οι κανόνες στα σημεία αυτά δεν θα μπορέσουμε να ορίσουμε δυστυχώς ε, πλήρως και είναι κρίμα γιατί εγώ πιστεύω ότι ε, στις προτάσεις, αν είχε επιτευχθεί συμφωνία για τις προτάσεις του, που είχαν υποβληθεί στον τρίλογο, στον τριμερή διάλογο, θα είχαμε, θα είχαμε κάνει ένα καλό βήμα μπρο. Όπω είπε και η Επίτροπο, αναγκαστικά θα πρέπει να το πάμε στην επόμενη θητεία. Κύριε Βίστινγκ, ένα 1,5 λεπτό. Η νομοθεσία που ψηφίζεται σήμερα σε ό,τι αφορά τι κοινωνικέ εισφορέ και τι κοινωνικέ παροχέ ε, στην Ευρώπη αποτελεί ένα λυπηρό ορόσημο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τη σχέση με το δανεικό μοντέλο. Πρόκειται για κοινωνικό τουρισμό, κοινωνικό dumping και ένα βήμα προ τη λάθο κατεύθυνση. Γιατί τα συστήματα κοινωνική ασφάλεια δεν θα σημαίνουν ίσα δικαιώματα για όλου του πολίτε. Η Ευρωπαϊκοί, οι Ευρωπαίοι πολίτε θα έχουν καλύτερη θέση, καλύτερη, ε, μεγαλύτερη προτίμηση σε σχέση με του εθνικού εργαζόμενου σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τι ε, συνεισφορέ. και νομίζω ότι είναι σημαντικό για μα να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε τα εθνικά συστήματα πρόνοια και θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι ίσοι οι όροι για όλου. και αν δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή των επιδομάτων, παροχών αυτών. Είτε μιλάμε για επιδόματα, είτε μιλάμε για άλλου είδου παροχέ, οι οποίε χορηγούνται σε Ευρωπαίου πολίτε στην Δανία. Ευχαριστώ, κύριε Τόμ, για 1,5 λεπτό. Η κυρία Τόμα, ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μία από τις τέσσερις ε, βασικές ελευθερίες είναι η ελεύθερη μετακίνηση και αυτό δεν είναι δυνατόν χωρίς ε, την ε, συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων. Όταν ε, έχουμε λοιπόν το θέμα αυτό, ένα από τους βασικούς λόγους ανησυχία μας είναι ότι μπορεί να χάσει κανείς τα δικαιώματά όταν ε, μετακομίσει σε άλλη χώρα. Και αυτό αποτελεί βασική ανησυχία των διασυνοριακών εργαζομένων σε ό,τι αφορά τον καλύτερο συντονισμό των ε, κοινωνικών συστημάτων. Δυστυχώ, λοιπόν είναι παροχημένη ε, η σημερινή νομοθεσία. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις Επιτροπές του Κοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις στο Συμβούλιο. Και αυτό σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι θα μας οδηγήσει σε μια κατακριματισμένη κατάσταση και στο μέλλον και θα ήθελα να σας πω ότι ο εθνικός, ε, οι εθνικές διακρίσεις των ε, εργαζομένων που μετακινούνται απαγορεύεται ρητά από τη συνθήκη. Θα ήθελα να πω και για τους ε, εργαζόμενους από τις ανατολικές χώρες και την πρόσβαση στις αγορές των δυτικών κρατών μελών ότι δεν είμαι υπέρ της προσαρμογής των επιδομάτων που θεωρώ ότι αποτελεί μια άδικη λύση η οποία οδηγεί σε μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος και θα πρέπει αυτό να μην συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κάρι, ένα λεπτό. Συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε ένα Θεμελιωδε ερώτημα σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδου ε, εθνικά θέματα. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ διαφορετικά μεταξύ του κοινωνικά συστήματα. Αυτό που είναι καλό για μια χώρα μπορεί να είναι καταστροφικό για μια άλλη. Πρέπει να προστατεύουμε του πολίτε μα χωρί να υποσκάπτουμε τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης. Η πρόταση την οποία συζητούμε σήμερα ενέχει αυτό το κίνδυνο να υποσκάψει το σύστημα της Δανίας το σύστημα της Δανίας βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης με τους ανέργους και μεταξύ των εργαζομένων. Η περίοδος των έξι μηνών είναι ένα σημαντικό θέμα και μπορεί να καταστρέψει το σύστημά μας δημιουργώντας κοινωνικό ντάμπινγκ. Είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει. Όχι πιστεύω. Ευχαριστώ. Για μισή λεπτό λόγο στην κυρία Ρέντκε. Thank you very much, Madam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επιτροπή, αξιότιμη συναδελφή. Το Brexit, το δράμα του Brexit, το οποίο εκτελήσεται στη Μεγάλη Βρετανία, θεωρώ ότι ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με το δημοψήφισμα. Εδώ και δεκαετίες έχουμε συστηματική ε, επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στη Μεγάλη Βρετανία. Και η συζήτηση αυτή έχει να κάνει και μια συζήτηση για την προσαρμογή των επιδομάτων. Μια συζήτηση η οποία δεν έχει να κάνει τίποτα και δεν συμβάλλει σε τίποτα στην κοινωνική δικαιοσύνη στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Μόνο δελτριάζεται την κοινή γνώμη. Θα ήθελα να πω το εξή. Η προσαρμογή των επιδομάτων τέκνου δεν θα λύσουν σε κανένα πρόβλημα. Δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα κοινωνική αδικία ούτε στη Μεγάλη Βρετανία ούτε σε άλλη χώρα. Ουσιαστικά θα δημιουργήσει μόνο μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν και αν θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά σε μια ενωμένη Ευρώπη, θα πρέπει να καταργήσουμε τέτοιε προσαρμογέ. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επίση ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Γιατί οι περιοχέ που πλήττονται από, αδικία, από κοινωνική αδικία και από φτώχεια είναι αυτέ που ψήφισαν αρνητικά στο δημοψήφισμα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι η προϋπόθεση για το Brexit υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά και την κοινωνική αειδικία το μίσος κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα εκρηκτικό μείγμα. Αν θέλουμε λοιπόν αυτό το κοινό ευρωπαϊκό έργο να αναπτυχθεί, θα πρέπει να το καταστήσουμε πιο κοινωνικό, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές και θέλουμε καλό συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων. Αυτό είναι απόλυτη προϋπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Επόμενη ομιλητρία για ένα μισή λεπτό, η κυρία zaapelować... Οι επόμενες διαπραγματεύσεις θα γίνουν από το νέο κοινοβούλιο και θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικό το νέο κοινοβούλιο, ιδίω ό,τι αφορά του τους μετακινούμενους Αυτοί που πηγαίνουν σε άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να καλύπτουν το συντομότερο δυνατό από τα κοινωνικά συστήματα τη χώρα υποδοχή. Η περίοδος ε, μπορεί να επεκταθεί αν έχουν ε, από τρει έξι μήνε αν χρειάζονται να ενταχθούν σε νέο σύστημα. Επίση, χρειάζονται λύσει για του μετα για τους διασυνοριακούς υπαλλήλους. Η τιμαριθμιμοποίηση είναι εκτός ε, συζήτησης. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα ήδη αντιμετωπίζουν μεγάλη γραφειοκρατία όσο έχει με βάση την απέτηση για την εξουσιοδότηση. Μπορείτε να πάτε λίγο λιγότερο γρήγορα. Ναι για να αποφύγουμε λύσεις κατά, με βάση τις οποίες το, η αγορά της κοινωνικής ασφάλισης θα ε, κατακαιρματιστεί. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια ως προς το ποιος καταβάλει και από πού ε, τα επιδόματα και από πού παρέχεται η κοινωνική ασφάλιση. Επίσης πρέπει η διατύπωση του άρθρου 13 του για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, όπως οι οδηγοί. Αυτοί πρέπει να καλύπτονται από την χώρα κατοικίας. Το νέο κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι οι νέοι συνάδελφοι θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Ο κύριος Πάβελ, ένα, λεπτά, ένα λεπτό. Πρόεδρε Πίτροπε, ευχαριστώ για την πρόταση και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζετε την τιμαριθμοποίηση. Και ευχαριστώ που δώσατε, δείξατε αποφασιστικότητα. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με την Αυστρία για τη διαδικασία παραπομπής θα παραταθεί στη συζήτηση αυτή κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να αποκαλούν τον εαυτό τους αριστερούς ξέχασαν τι σημαίνει κοινωνικό dumping και τι σημαίνει ίση αμοιβή για αντίστοιχη δουλειά. Αυτό σημαίνει και ισότιμη ε, αντιμετώπιση όλων των Ευρωπαίων. Να μην χάνουμε ψήφους προς όφελος της άκρας δεξιάς. Η έκθεση αυτή προφανώς είναι μια συμβιβαστική λύση, προωθεί ωστόσο την Ευρώπη και πρέπει να περάσει. Ευχαριστώ. Thank you for one minute, Madam ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διακίνηση των εργαζομένων άνοιξε το θέμα τη κοινωνική ασφάλιση των διαμεθοριακών εργαζομένων. Για να μπορούν να υποφελούνται των δικαιωμάτων του, οι μεθοριακοί εργαζόμενοι ε, θα αναγκάζουν τα κράτη-μέλη να συντονίζονται καλύτερα και να ε, ευθυγραμμίσουν τις νομοθεσίες τους. Είναι προφανές ότι χρειάζονται βελτιώσεις σε αυτό το τομέα. Όμως δεν μπορώ να δεχτώ την προτινόμενη λύση γιατί εισάγει πιο περίπλοκους κανόνες και ανοίγει καινούριου ορίζοντες στην απάτη. Στους ε, ε, οι παροχές, οι κοινωνικές παροχές, οι μετακινούμενους εργαζόμενους θα πρέπει να πληρώνονται από το κράτος μέλος προέλευσης. Μπαίνοντα στην αγορά εργασία σε ένα άλλο κράτο μέλο, θα πρέπει ο εργαζόμενο να χάνει το δικαίωμα παροχών στο κράτο μέλο προέλευση ή στο κράτο μέλο ε, στο οποίο ε, ασκούσε προηγουμένω το δικαίωμά του περισσότερο, πιο περίπλοκες διατάξεις ε, μπορεί να δείχνουν πιο ωφέλιμες για τους εργαζόμενους, αλλά δημιουργήσουν μεγάλο βάρος στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ευχαριστώ. Γκάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο κόμμα μου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί όμως αυτό ο στόχο με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, γιατί δημιουργεί νομική ασφάλεια. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα εξαιτία των διαφορών μεταξύ ε, ε, εργαζομένων. Θα γίνει εξαγωγή παροχών. Οι προτάσεις οποίες εμείς ε, υποστηρίζουμε δυστυχώς δεν εγκρίθηκαν και δεν πέρασαν στο τελικό κείμενο. Θα προτιμούσαμε προφανώς, φαντάζομαι, την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Θα καταψηφίσουμε το κείμενο όπως έχει προταθεί ένα Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφορετικά συστήματα κοινωνική ασφάλιση, διαφορετικού κανόνε, προπολογισμού και κανόνε για το πώ κατανέμει τα επιδόματα ανεργία, μητρότητα, πατρότητα, τα οικογενειακά ή προσύνταξοδοτικά επιδόματα. Όμω, όσα επιδόματα και αν μπαίνουν, τα ερωτήματα είναι αμέλικτα. θέλουμε ή δεν θέλουμε μια νέα ευρώπη θέλουμε ή δεν θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων; θέλουμε ή δεν θέλουμε να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των Δανού ή των Έλληνα εργαζομένων όταν αλλάζει τόπο διαμονής. στηρίζουμε την έκθεση μπάλας που υποστηρίχθηκε και από ένα ευρύ φάσμα βουλευτών. μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε νέο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό σύστημα. αυτός είναι και ο δρόμος για νέο φορολογικό σύστημα χωρίς διαφορές μεταξύ μας για να χτίσουμε μια πραγματικά ενωμένη ευρώπη. Λόπες Φοντανιέ, για ένα λεπτό. Εμεί εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύεται από την εγγύηση των δικαιωμάτων του. Είναι κρίμα που δεν εξασφαλίστηκε ε, η κατάλληλη η σχετική πλειοψηφία στο Συμβούλιο γιατί οι προτάσει είχαν πολλές, θετικ... πολλές θετικές πλευρές. Ε, που θα ενίσχυαν την ελεύθερη κυκλοφορία. Ο συντονισμός ε, των, ε, της μακρόχρονης Περίθαλψη, καθώς επίσης και η, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή ήταν πολύ θετικέ πτυχές. Ε, θέλω να πω ότι μια και είναι η τελευταία μου παρέμβαση εδώ στο Κοινοβούλιο θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω ευχαριστώντα σας για τα τελευταία δέκα χρόνια. Εργαστήκαμε πολύ με συνένεση μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών ομάδων ιδιαίτερα στην Επιτροπή Απασχόλησης, ε, κάναμε μια πολύ καλή δουλειά ε, για τους λιγότερο ευνοημένους. Είναι μια προσπάθεια η οποία πολλές φορές είναι άγνωστη στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ελπίζω και εύχομαι αυτή η συνένεση να συνεχίσει να υπάρχει και στην επόμενη θητεία γιατί είναι πολύ σημαντική για να καταφέρουμε μια πιο ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και την Επίτροπο. Ευχαριστούμε και την κυρία Λαπεφοντανιέ και είμαι βέβαιη ότι το κοινό θα ενημερωθεί για τη δουλειά του Κοινοβουλίου εγκαίρως. Ο κύριος Τέτιαν για ένα λεπτό έχει το λόγο. Αξιότιμη Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, σήμερα θα είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια επιτυχία σε ό,τι αφορά και την οδηγία για την απόσπαση, ή διαργασία ίδιος μισθός, ίδια δικαιώματα κοινωνικά στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε ως Ευρωπαίοι και αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε ως λάβαρο. Κάναμε μια καλή πρόταση η Ευρωπαϊκή ενιαία Αγορά δεν αποτελεί μόνο από το ευρώ και από την ελεύθερη μετακίνηση, αλλά και από κοινωνική ασφάλιση για τα δικαιώματα αυτά. Τα δικαιώματα τα οποία προβλέπετε στο κείμενο του κ. Μπαλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την κινητικότητα των ανθρώπων και πρέπει να υποστηρίξουμε του εργαζόμενου σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των επιδομάτων και των παροχών. Δεν έχουν οποιαδήποτε τεκμηριωμένη βάση. Γεγονό είναι ότι υπάρχει εθνικιστική προπαγάνδα γιατί δεν είναι χιλιάδε οι άνθρωποι που θα κάνουν τέτοιες καταχρήσεις. Αύριο θα ψηφίσω υπέρ της αναθεώρησης ε, των γενικών συστημάτων, γιατί αυτά, το παιχνίδι μεταξύ ανατολή και Δύση σε Βορρά και Νότου, αυτό ας το αφήσουμε στους εθνικιστές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φοντεκάν Λάρα για ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, χτες ε, εγκρίναμε την ε, δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας σε ό,τι αφορά και τις συμβάσεις, τις εργασίας, ε, τις συμβάσεις ε, απόσπασης, σε ό,τι αφορά την ίδια εργασία και την ίδια μισθό και σε ό,τι αφορά την ισορροπία οικογενειακού και εργατικού βίου. Επίση, η, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το κοινωνικό τη πρόσωπο. Βλέπουμε όμω ότι το συγκεκριμένο τεχνικό θέμα έχει μεταφραστεί σε ένα εκρηκτικό μείγμα στον τύπο. Και πρέπει να αποφασίσουμε τελικά ποιο κράτο είναι υπεύθυνο για την παροχή επιδομάτων και το πώ κινούνται οι άνθρωποι μεταξύ των πτυχών του κοινωνικού ιστού. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, Έχουμε εργαζόμενου ε, από το Βέλγιο που πήγαν στη Γερμανία και διαπιστώσαν τελικά ότι δεν έχουν ε, δικαίωμα σε ε, επιδόματα ανεργία ούτε από το Βέλγιο ούτε τη Γερμανία. Δεν συμφωνώ με την πρόταση ενό μήνα για το παροχή δικαιωμάτου ανεργία. Συμφωνώ με την πρόταση τη κυρία Τέισεν, γιατί με ένα μήνα δεν θεωρώ ότι μπορεί κανεί να έχει εργασιακή σχέση Συχνά μιλάμε για τουρισμό ε, σε ό,τι αφορά τα κράτη τη κοινωνική πρόνοια, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήθελα να το έχω αναφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κρίστενσεν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Επίσης, συμφωνώ να δώσουμε ασφάλεια στους εργαζόμενους. Χρειαζόμαστε όμως μια καλύτερη ισορροπία από αυτή που έχει τώρα η έκθεση Χρειαζόμαστε σωστά δικαιώματα και μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει διάκριση εις βάρος των ημεδαπών εργαζομένων σε σχέση με τους αλλοδαπούς. Αυτό πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά εργασίας έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ανέργων για μικρό χρονικό διάστημα. Η χώρα προέλευση του εργαζομένου έχει μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την περίπτωση, άρα χρειαζόμαστε μια περίοδο μακρύτερη από τους τρει μήνες. Έξι μήνες προτάθηκαν. Έχουμε διαφορετικές πολιτικές ε, αγοράς εργασίας και διαφορετικές επιπτώσεις από αυτή τη νομοθεσία. Υπάρχει ωστόσο και το πρόβλημα της εξαγωγής των ε, επιδομάτων. Εμείς θεωρούμε ότι η αρχή της εξαγωγής των τριών μηνών πρέπει να παραμείνει. Σε ό,τι αφορά τους μεθοριακούς εργαζομένους, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη σαφήνεια από ό,τι παρέχει το σύστημα τώρα. Ο κ. Λένας. ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ζουν και εργάζονται σε άλλα κράτη-μέλη εκτό από το κράτο προέλευσή του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να έχουν κοινωνική πρόνοια. Δεν μπορεί κανεί να είναι θύμα πολύ απλά επειδή περνάει τα σύνορα και κυρίως όταν ε, ζει κανείς σε μια μεθοριακή περιοχή όπως το δικό μου Λιμβούργο και παρόλα αυτά θα καταψηφίσω αυτό το κείμενο που ρυθμίζει πάρα πολύ καλά πράγματα με πόνο καρδιά ε, και κυρίω ε, λόγω των ε, επιδομάτων ανεργία. Είναι σημαντικό το επίδομα ανεργία και όποιο χάνει τη δουλειά του θα πρέπει να βρίσκει γρήγορα δουλειά. Αυτό είναι καλό και για το άτομο αλλά και για την κοινωνία, για όλου μα λοιπόν. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή κίνητρα λοιπόν, πραγματικά κίνητρα για να ψάχνει κανεί ενεργά για θέσει απασχόληση. Και βλέπουμε ότι αυτά τα κίνητρα πραγματικά υπονομεύονται από τον τουρισμό επιδομάτων. Στην Ολλανδία έχουμε 4.000 τέτοια επιδόματα ανεργία τα οποία εξάγονται. Από τα 4.000 αυτά επιδόματα, 0,6% βρίσκει θέση απασχόληση κατά τη διάρκεια ισχύω του επιδόματο ανεργία. Αυτό πραγματικά είναι υπερβολικά μικρό ποσοστό, γελία μικρό ποσοστό. Και χρειαζόμαστε λοιπόν κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό υπονομεύει όμω την αίσθηση δικαιοσύνη στην κοινωνία μα. Και τώρα θέλουμε να διπλασιάσουμε την περίοδο. Αμα εξαγωγή των επιδομάτων χωρί να προσθέσουμε οποιοδήποτε κίνητρο για την εξέφραση εργασία. Αυτό πραγματικά είναι παράλογο, απαράδεκτο για την ΣΕΝΤΕΑ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for one minute, Madam Arena. Arena, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ των οποίων και η ελευθερία κυκλοφορία, συνοδεύονται από κανόνε. Οι κανόνες για την κινητικότητα των εργαζομένων είναι κανόνες κοινωνικής προστασίας, διότι η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη κοινωνικής προστασίας. Είναι όμως και κανόνες μια θέμη του ανταγωνισμού. Η αναθεώρηση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως προτείνει η έκθεση του συναδέλφου Μπάλας, πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι βέβαια τέλεια αναθεώρηση, αλλά υποβάλει σαφείς προτάσεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ένωση και για να καταπολεμήσουμε την απάτη που ασκείται όχι από τους άνεργους που πηγαίνουν να κάθονται στον ήλιο και να ξεκουράζονται, αλλά από ε, ε επιχειρήσεις που θέλουν να μην προστατεύουν τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν πρέπει να πολεμήσουμε αυτόν, το, αυτή τη μορφή του αθέμητου ανταγωνισμού και πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση για να επιβεβαιώσουμε μια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι θέση της Ένωσης, ευρωπαϊκή θέση και να μην υποστηρίξουμε εθνικές ή εθνικιστικές θέσεις κάποιων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό η κυρία Ριμπέιρο. Αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λόγο θα ήθελα να κάνω ένα απολογισμό των προτεραιοτήτων. Αυτή η πρόταση καταδεικνύει τις κοινωνικές προτεραιότητες τις οποίες έχουμε υποστηρίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών η προστασία των, του κοινωνικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μοναδικό στον κόσμο. Προστατεύει τους πολίτες σε όλες τις φάσεις ζωής τους, εγγυάται καλύτερη αξιοπρέπεια, βελτιώ, καλύτερες ε, κοινωνικές συνθήκες, ε, σύγκληση, κοινωνική σύγκληση, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη. Μια Ευρώπη οποία αποφελείται της κινητικότητας, της διαφορετικότητας, της ποικιλομορφίας της ε, και των διαφορετικών εκατοτήτων κάθε πολίτη. Η κινητικότητα θα πρέπει να συνδέεται με μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη για να μην τύχαν εκμετάλλευσης οι ευάλωτοι εργαζόμενοι. Η Ευρώπη μετά όμως ε, δεν πρέπει να βρίσκει καταφύγιο στους εθνικισμούς. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη τα ε, οποία ε, χρησιμοποιούν και υποφελούνται των γνώσεων των μετακινούμενων εργαζομένων και των αποσπαζόμενων εργαζομένων θα πρέπει να τους στηρίξουν και με, τα, με κοινωνικά επιδόματα. Τα κοινωνικά επιδόματα θα πρέπει να πληρώνονται στο επίπεδο, στο ύψος των επιδομάτων του, της χώρας στην οποία εργάζονται οι εργαζόμενοι. Εκεί θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ντόπιου εργαζόμενους. Η ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να συνδέεται με την προστασία για μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο ίση. Ήταν τιμή μου να εκπροσωπώ τους Πορτογάλους εδώ και ελπίζω η κληρονομιά ε, ε, να είναι μια Ευρώπη πιο κοινωνική. Ευχαριστώ. να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συνεισφορά σας και τις συμβολές σας. Ε, εργαστήκαμε πάρα πολύ καλά στην Επιτροπή Γεωργίας και σας εύχομαι ότι καλύτερο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σμόλκοβα τώρα είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη κινητικότητα των ατόμων, των εργαζομένων, των υπηρεσιών και είτε πρόκειται για αναψυχή, είτε πρόκειται για εργασία και αντιμετωπίζουμε λοιπόν το θέμα αυτό με τις ε, διασυνοριακέ. Ε, περιοχές και τους ε, εργαζόμενους. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό χωρίς ε, γραφειοκρατία. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα θέματα της γλώσσας, ε, τα θέματα των λοιπόν εμποδίων. Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό έργο το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, χωρί διαφορά, έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συντονισμό θα πρέπει να συζητηθεί επί της αρχής, γιατί κάποια κράτη-μέλη σήμερα, σήμερα ήδη προσαρμόζουν τα επιδοτήματα, τα, τα επιδόματα οικογενειακά. Και έτσι αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση για τους εργαζόμενους από άλλα κράτη-μέλη. Ένα αρνητικό παράδειγμα είναι η Αυστρία με την προσαρμογή των επιδομάτων τέκνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάμικινς έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αύξηση της κινητικότητας σημαίνει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να τύχουν καλύτερης προστασίας. Ωστόσο, αυτό πλοκάρεται από μια μειονότητα, μια ψηφία στο Συμβούλιο. Μιλάμε όμως για θέματα τα οποία είναι ύψης της σημασίας για τους εργαζόμενους, τα θέματα από κοινωνικών παροχών. Και αυτό επηρεάζει και το πώς ε, αντιλαμβάνονται οι πολίτες την ποιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν δίνει τέτοια σημασία στα κοινωνικά επιτόματα, στις κοινωνικές παροχές. Κάποιες χώρες φαίνεται ότι θέλουν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό βάζει τα κοινωνικά μας συστήματα σε ανταγωνισμό. Και όντω, στο τρέχον πλαίσιο, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν για τις κοινωνικές παροχές. Αλλά οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ε, αρχή της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόμπερν, μισή λεπτά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Ωραία όλα αυτά. Αυτό όμως είναι πολύ επικίνδυνο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινωνική προστασία στηρίζεται ε, στις ανάγκες, όχι στις εισφορές όπως την Ήπειρο. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, μπορεί να εισπράξεις μόνο ό,τι έχεις καταβάλει στο σύστημα. Αν δεν έχεις ε, καταβάλει, δεν εισπράττεις. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο, κυρίες και κύριοι, σπρώχνονται στο καλέ οι μετανάστες για να έρθουν στη Βρετανία και δεν σπρώχνονται στο Ντόβερ για να έρθουν στη Γαλλία. Γιατί στη Βρετανία το, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ πιο ανοιχτό στους νέους εισερχόμενους. Αυτό δεν είναι κακό. Ε, το πρόβλημα είναι ότι και τα δύο συστήματα έχουν υπέρ και κατά, αλλά μεταξύ τους είναι ασύμβατα. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα αυτό θα οδηγήσει σε κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της Βρετανίας. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που υπερψηφίσαμε το Brexit. Μας ανησυχεί το ότι θα διαλυθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και θα υπάρξει τεράστια ποιήση στο, σύστημα, στο εθνικό σύστημα υγείας. Θα έρθουν όλοι και θα χρησιμοποιούν το σύστημα.